Bonjour à tous, nous allons commencer notre... Καλημέρα σα θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Καταρχάς, έγκριση της μερίσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια για το σχέδιο της μερίσιας διάταξης. Όχι, επομένω εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Στην συνεχεία έχουμε για ένα λεπτό την ώρα των ερωτήσεων. Δεν έχω λάβει ε, κάποια ερώτηση για την Επιτροπή σήμερα. Άρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ούτε ανακοινώσει έχω. Αντικαθιστώ την Εύα γιατί είναι σε αποστολή στην Σενεγάλη. Σήμερα δεν έχω κάποια ανακοίνωση να σας κάνω, άρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να μας αναγγείλει κάτι. Όχι, από ό,τι βλέπω. Ωραία. Σημείο 5, λοιπόν, η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΑΦΕΤ για τις εκλογές ε, στο Νότιο Σουδάν. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της αντιπροσωπείας ε, παρατήρησης των εκλογών. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που συμμετέχετε στην κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών ανάπτυξη εξωτερικών για τις εκλογές στον Νότιο Σουδάν. Ο συνάδελφος ε, Ιωάννα Μίρτσα Πάσκου, αν το προφέρω σωστά το όνομά σας, από την Επιτροπή Εξωτερικών είναι εδώ μαζί μας, τον καλωσορίζουμε. Θα θυμάστε ότι προσφάτως η Επιτροπή Ανάπτυξης και η Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, διοργάνωσαν μια κοινή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν μετά το δημοψήφισμα με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ε, των ε, προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν. Σήμερα ουσιαστικά έχουμε διαφορετικούς στόχους θέλουμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον εισηγητή μας που θα μας εκθέσει την ε, αναφορά της αντιπροσωπείας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την αποστολή παρατήρησης των εκλογών. Θα γίνει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ε, του δημοψηφίσματος και θα δούμε ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις από τις διαπραγματεύσεις που ακολουθούν τις εκλογές. Καλώς ορίζω λοιπόν τους ομιλητές μας την Μαριάν πρώτα απ' όλα που ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικής Παρατήρησης. Η κυρία Βερονίκ Τεκάιζερ, συνάδελφός μας, δεν μπορεί να έρθει ότι ασθενή. Η κυρία Ρόζαλιν Μάρσιν που είναι ειδική εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου για το Σουδάν είναι επίσης μαζί μας. Ο κύριο Αμασούρ Εμπρέμ Μπολάμ Δουρντάιν, πρέσβη του Σουδάν στι Βρυξέλλες, εξοχώτης λοιπόν ο πρέσβη είναι εδώ και ζητώ συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ο κύριο Ναζάριο από το γραφείο σύνδεση της ε, ε, του Νοτιού Σουδάν. Η συνάδελφό μα, η Μαρία, η Μαρία Νεντέλη, θα έχει διάθεση 10 λεπτά για να μας ε, εκθέσει την αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και κάθε ομιλητής ε, που θα ακολουθήσει θα έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Θα έχουμε στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων με τους ε, βουλευτές, αλλά πριν δώσω το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί υπάρχει μια βαθιά δέσμευση ε, του πληθυσμού του Νοτίου Σουδάν, που αποφάσισε να επιλέξει το πεπρωμένο του είναι σημαντικό το λιθαράκι που μπήκε, πιστεύω, με, την, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, γενικότερα για την ειρήνευση στην περιοχή. Τα αποτελέσματα του δημοψήφισματος δεν ξέρω αν τα έχουμε. Τα έχουμε. Δεν τα έχουμε ακόμη αυτή τη στιγμή, άρα δεν μπορώ και να σας τα παρουσιάσω. Καλούμε λοιπόν χωρίς καθυστέρηση από όλες τις πλευρές να επιληθούν όλα τα ζητήματα ώστε να έχουμε την Γενική Συμφωνία Ειρήνευσης και πρέπει να λυθούν βέβαια και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά με σεβασμό ε, στην ε, ελευθερία και τα δημοκρατικιώματα του λαού του Σουδάν. Επίσης, θέλω να εκφράσω τη βαθιά ανησυχία μου ενώπιση της κατάστασης στην περιοχή Αμπιέ. Υπάρχουν ε, βία επεισόδια και στην περιοχή του Νταρφούρ. Έχουμε 40.000 νέους εκτοπιστέντες και υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζει και η ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου. Θα δώσω όμως τώρα το λόγο στην ε, κυρία Νεντέλσεβα. Μαρία, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης και της ΑΦΕΤ, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μπορώ να μοιραστώ ε, μαζί σας τις εντυπώσεις, τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαρτιζόταν από έξι μέλη που ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό τους, τη δέσμευση και την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς. Ευχαριστώ την κυρία Ντεκάιζερ για την εξαιρετική συνεργασία και την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αποστολή παρατήρησης των εκλογών και στο Χαρτούμ και στη Τζούμπα. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη της Γραμματείας, χωρίς την οποία αυτή η αποστολή δεν θα στεφόταν από επιτυχία. Η παρέμβασή μου θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Καταρχήν θα σταθώ στην ίδια την εκλογική διαδικασία, όπως είχε επιτοπίως και μετά θα μιλήσω για τις πολιτικές προκλήσεις που διαγράφονται κατά την ψηφοφορία. Ως προς την διεξαγωγή των εκλογών μπορώ να πω ότι ήταν ειρηνική διαδικασία και πολύ καλά οργανωμένη. Αν και έφτασαν ανισχυτικά μηνύματα πριν από δύο-τρεις μήνες διαπιστώσαμε ότι κατά την διεξαγωγή των εκλογών δεν είχαμε μείζωνα ατυχή περιστατικά. Και αυτό ε, βεβαίως μας δείχνει ότι θα πρέπει να καταβάλουμε και άλλες προσπάθειες. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή Διενέργειας των Εκλογών και στο Βόρειο και στο Νότιο Σούδαν. Πριν μιλήσω για τις εκλογικές περιφέρειες που ήταν σε, είχαν πολύ καλό επίπεδο και στο Χαρτούμ και στη Τζούμπα, καθώς και στην περιοχή της Τερεκέκα που επισκεφθήκαμε για να δούμε πώς διεξάγεται η ψηφοφορία. Κατά τη ε, διάρκεια της διεξαγωγής είχαμε επαφές με την κεντρική αποστολή παρατηρήσεις, επίσης τακτική ενημέρωση από την επικεφαλή στην κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ και από τους εμπειρογνώμονες που μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Πιστεύουμε ότι γι' αυτό ακριβώς επέτυχε και η αποστολή μας. Τώρα, σε σχέση με τις πολιτικές ε, προκλήσεις, αλλά και οικονομικές και κοινωνικές, διότι είναι αλληλένδετες, θα πρέπει να υπογραμμιστούν πολλά στοιχεία. Θα μπορούσαμε να δούμε τις προκλήσεις για το βορρά ή το νότο και για τις προκλήσεις, τις κοινέ προκλήσεις και των δύο χωρών. Ως προς τις προκλήσεις για το βορρά, τίθεται το θέμα της τήρησης των αποτελεσμάτων από τις αρχές του Χαρτούμ, που θα είναι η βάση για τις ε, μελλοντικές ε, διαπραγματεύσεις της 9 Ιουλίου, όπου θα επικυρωθεί η ανεξαρτησία. Επίσης θα πρέπει να ανοίξει ένας πολιτικός χώρος. Οι αρχές του Χαρτούμ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα νέα δεδομένα με βάση τον πολιτικό πλουραλισμό έτσι ώστε να δεχτούν την πολιτική, θρησκευτική και εθνοτική διαφοροποίηση για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Υπάρχουν πολλά εκρεμή ζητήματα ως προς το Νταρφούλ, αλλά επειδή η αποστολή δεν βρέθηκε επιτόπου, δεν θα ήθελα να σταθώ στις λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ασφάλεια εκείνων που ασχολούνται με ανθρωπιστικά ζητήματα είναι μείζονος σημασίας. Ως προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την υπόθεση Αλμπασίρ δεν μπορούμε να την παραλείψουμε εδώ. Για τις προκλήσεις του Νοτίου Σουδάν οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις και η δημιουργία μιας μεταβατικής κυβέρνησης μας απασχόλησε και θα παρακολουθήσουμε εκ του και στη διαδικασία ως προς τον πολιτικό πλουραλισμό και αυτό είναι μείζον σημασία. Το SPLM ως απελευθερητικό κίνημα δεν θα πρέπει να έχει αποκλειστικό ηγετικό ρόλο. Επίσης, η οριοθέτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων των ενόπλων δυνάμεων και των κομμάτων θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος. Κατά το δημοψήφισμα είδαμε ότι άμεσα τίθεται το θέμα των εκτοπισμένων ή των παλινοστούντων, δηλαδή εκείνο που εγκατέλειψαν το βορρά για να πάνε στο νότο. Ίσως ε, τους εκπλήξει η ζωή όταν επανέλθουν. Πρόκειται για νέα δεδομένα σε σχέση με την ηθαγένεια, αλλά αυτό ισχύει και για το Βορρά. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, πώς το νέο κράτος του Νότου θα μπορέσει να ε, ενσωματώσει όλους αυτούς τους πολίτες. Σε σχέση με αυτά που προελέχθησαν, μπορούμε να δούμε ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν ορισμένες κοινέ προκλήσεις. Το θέμα των συνόρων είναι επίγον. Θα πρέπει να εξευρεθεί μια λύση έτσι ώστε να μην ανακύψουν ε, συγκρούσεις. Επίσης, ε, οι ε, διάφορες συμπλοκές έγιναν ακριβώς σε αυτή την περιοχή. Ως προς το άνοιγμα του πολιτικού χώρου, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πλουραλιστικός πολιτικός χώρος όπου να υπερισχύει το κράτος δικαίου καθώς και οι θρησκευτικές και εθνοτικές ελευθερίες. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ειρηνική ατμόσφαιρα όπως είδαμε κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να συνεχιστούν γιατί τα δύο αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα. Ακριβώς επειδή είναι αλληλένδετα θα πρέπει να σταθούμε και σε δύο άλλα ζητήματα. Αφενός το θέμα του πετρελαίου και αφετέρου το θέμα του χρέους. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε αναπτυξιακά σχέδια και στις δύο χώρες. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό χώρο. Η ειρήνη και η σταθερότητα θα πρέπει να εξασφαλιστούν έτσι ώστε τα έσοδα από το πετρέλαιο να είναι υπέρ του, του ντόπιου πληθυσμού. Βεβαίως ζήσαμε μια ιστορική στιγμή. Διενεργήθηκαν πολύ καλά οι εκλογές, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις αμέσως μετά το δημοψήφισμα και πώς μπορούμε να άρουμε τα προσκόμματα. Αυτό έχει σχέση με την οικονομικοπολιτική και κοινωνική κατάσταση των δύο χωρών, θα πρέπει και οι δύο χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειες διαλόγου και συνεργασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει παρούσα και να συνεχίσει τις ε, σχέσεις και με τις δύο χώρες. Τέλος, ίσως είναι κάπως πρόωρο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στάση των 27 κρατών μελών. Πιστεύω ότι η αναγνώριση των δύο κρατών δεν θα πρέπει να γίνει ένας αγώνας δρόμου ανάλογα με τα κράτη. Θα πρέπει η Ευρώπη να μιλήσει με μία φωνή και επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το δημοψήφισμα του Σουδάν είναι το πρώτο που διενεργήθηκε μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Ροζαλίν Μάρτσεν. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα και με σημερινή συζήτηση για το δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν είναι πολύ επίκαιρη για τα τελικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος θα ανακοινωθούν στο Χαρτούμ ε, σήμερα το απόγευμα στις 5.30 ώρα Βρυξελών, για να είμαι πιο ακριβής, σε μια εκδήλωση που θα παρίστανται και ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός και αναμένεται να επιβεβαιωθούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δείχνουν ότι είναι 99,8% υπέρ της ε, ε, απόσχησης. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την ειρνευτική διαδικασία σε ό,τι αφορά και την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενεί τις Σουδανικές Αρχές για την διοργάνωση του δημοψηφίσματος παρά από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και συμμετείχε συντριπτική πλειοψηφία των καταχωρισμένων ε, ε, ατόμων για να εκφράσουν την επιθυμία τους για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Πρόκειται για ένα σουδανικό επίτευγμα βασικά, αλλά και μια επιτυχία της ε, εθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αφρικανικής κοινότητας και του αφρικανικού πάνελ, του οποίου προεδρεύει ο πρόεδρος Μπέκη των Ηνωμένων Εθνών, της, των ΙΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σουδάν ήταν σε υψηλή θέση ε, στις συζητήσεις των Υπουργικών Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο, Νοέμβριο και την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκαν αυτά από τους Υπουργούς Εξωτερικών ε, τονίζοντας τη σημασία που έχει να βρεθεί να καταφέρουμε να διοργανώσουμε ένα ε, επίκαιρο δημοψήφισμα το οποίο το αποτέλεσμα θα γίνει σεβαστό από όλους και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του τελευταίου Σεπτεμβρίου και της συνεδρίασης με τον Μπάκι Μουν και διαφόρων άλλων συναντήσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και εγώ επανέλαβα σε όλες μου τις επαφές τα μηνύματα αυτά, σε όλες μου τις επαφές με τις Σουδανικές αρχές και άρα υπήρχε υψηλή ε, διπλωματική δέσμευση σε όλο τον κόσμο η αποστολή μιας εξειδικευμένης αποστολής παρατήρησης τη Σουδάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και αύξησε επίσης την πολιτική σημασία της Ένωσης. Στη συζήτηση στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα, η πρώτος εκπρόσωπος ε, ευχαρίστησε την κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ και την ομάδα της στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σημασία και το ρόλο που έπαιξαν για να δημιουργηθεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνη προς το δημοψήφισμα και θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω την κυρία Βερονίκ Δικάιζερ και την κυρία Μαρία Ντατζέβα για την ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρηματοδότηση και τεχνική αρρωγή για να υποστηρίξει τις αρχές της Σουδανικές για την εξάγωγη του δημοψηφίσματος αναμένοντα τα αποτελέσματα, τα βελικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως θα σεβαστεί τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ως αποτύπωμα, αν θέλετε, του πραγματικ της πραγματικής του Σουδανικού λαού και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανυπομονεί να εμβαθύνει την εταιρική σχέση με το Νότιο Σουδάν που θα καταστεί κατά πάσα πιθανότητα ε, νέο ναι, ανεξάρτητο κράτος μόλις ε, ε, καταγγελθεί η τρέχουσα σύμβαση τον Ιούλιο του 2011. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης του Νοτιού Σουδάν. Συγγνώμη, λέει η Αμιλήτρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει την προθυμία της κυβέρνησης του Σουδάν να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και στην πρωτεύουσα Τζούντα επιβεβαιώθηκαν αυτά καθώς και σε μια συνευρία στην Αντισαμπέμπα. Επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος από την κυβέρνηση του Σουδάν. Παρά το γεγονός ότι το δημοψήφισμα στέφθηκε με επιτυχία. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μωρών για να, φτάσει, να φτάσουν σε μια καλή συμφωνία για όλα τα θέματα και τα βασικά ζητήματα που θα προκύψουν στις σχέσεις μεταξύ Νότιου και Βορείου Σουδάν. Η περιοχή MBA εξακολουθεί να αποτελεί βασική, βασικό, βασική αιτία ανησυχίας και θα καλέσουμε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την του ουσιώδους λύσης για να βρεθούν και να στεθούν τα σωστά θεμέλια για τις μετέπειτα σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Επίσης, θα συνεχίσουν οι διαβουλέψεις και χαιρόμαστε που που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο γαλάζιο νήλο. Θα τεθούν θέματα ιδιαίτερα υπηκότητας, ασφάλειας, ε, ε, κοινή διάθεσης των εσόδων και καλώς μα μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει επί των βασικών αρχών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη δύο κρατών με κοινά σύνορα. Αλλά φυσικά πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για συγκεκριμένα θέματα. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πρόεδρου Μπέκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, παρέχει, παράσχει ε, χρηματοδότηση και τεχνική αρρωγή προς την ομάδα του κυρίου του Πέντρο Μπέκη, αξιότιμοι βουλευτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δεσμεύεται για την υποστήριξη και του Νοτίου και του Βορείου Σουδάν για την, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτου δικαίου και μια ε, ειρηνική, ενό ειρηνικού μέλλοντο για τον λαό του Σουδάν. Θα συνεχίσουν λοιπόν και θα ενισχυθούν ε, από πλευρά Ένωση ε, ο διάλογο και, με το με Βόρειο και με το Νότιο Σουδάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη δεσμευμένη για να παρέχει βοήθεια σε άτομα που πλήττονται σε περιοχές εμπόλεμες, στον Ταρφούρ, στο Νότιο Σουδάν. Επίσης, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δηλώσει ότι θα εξετάσουν την παροχή βοήθειας προς το Σουδάν σε ό,τι αφορά το, το χρέος του Σουδάν. Και στο Νότιο Σουδάν θα υπάρχει διαρκής αρρωγή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα γεωργίας, βασικών ε, υπηρεσιών κοινή ωφελία και μακροπρόθεσμα θα συνεχιστεί η αρρωγή μας. Αύριο θα μεταβώ στο Σουδάν με μια αποστολή τεχνικών εμπειρογνωμόνων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αξιολογήσουν τη μελλοντική συμβολή της Ένωσης στο Σουδάν και αν και σήμερα η συζήτηση εστιάζεται στο Νότιο Σουδάν, να μην ξεχνάμε το Νταρφούρ, το οποίο πρέπει να λαμβάνει διεθνή προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για τα περιστατικά βίας στο Νταρφούρ και ζητούμε από όλες τις πλευρές να διακόψουν τις ε, εχθρικές πράξεις και να εξεύρουν μια πολιτική λύση. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για, στα πλαίσια του γύρου της Ντόχα και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να βρεθεί η λύση. Και εξακολουθούμε να καλούμε την κυβέρνηση του Σουδάν να συνεργάζεται με το Διεθνές Δικαστήριο. Πρέπει να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης γιατί θα καθυστερήσουμε και έτσι θα χάσει χρόνο και η συνέντευξη των συντονιστών που ακολουθεί. Πρέπει να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Μετά τις 19 Ιουλίου θα υπάρξουν δύο κράτη στο Σουδάν και καθένα εξ αυτών θα χρειάζεται νέο σύνταγμα. Και στη Ζούντα και στο Χαρτούμ γίνεται συζήτηση για να αποταθεί χείρα προς τους εχθρούς. Πρόκειται για μια ευκαιρία και είναι τεράστιος ο ρόλος που μπορεί να διδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ε, ειρηνικό μέλλον για το Σουδάν και στο βορρά και στο νότο για να συνδράμει στους λαούς αυτούς σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά θέλω να υπενθυμίσω σε όλους τους ομιλητές να σέβεστε το χρόνο αγόρασης, παρακαλώ, γιατί πάντοτε έχουμε προβλήματα στις συνεδριάσεις μας. Πέντε λεπτά σας παρακάλεσα. Σας παρακαλώ σεβαστείτε και το έργο των υπολείπων. Εξοχότατος, αυτό εξοχότης ο πρέσβης τώρα παρακαλώ έχει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης που με προσκάλεσε να συμμετάσχω στη συνεδρία αυτή. Είμαι στην πρεσβεία λοιπόν του Σουδάν στη... στις Βρυξέλλες. Θέλω να ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας και πρέπει να πω ότι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την περίοδο και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εκ των προτέρων για την βοήθεια που θα παράσχετε και στο μέλλον ε, στη χώρα μας. Ασκήσαμε τον Ιανουάριο το δικαίωμά μας στο πλαίσιο της Γενικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας και αποφασίσαμε να ε, συγκροτήσουμε το δικό μας ανεξάρτητο ε, κράτος. Η κυβέρνηση εξέφρασε την πρόθεσή της να σεβαστεί την απόφαση και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την επίλυση των εκκρεμωτήτων. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται τα σύνορα, η ηθαγένεια, το νερό, το νόμισμα και βέβαια το ζήτημα της περιοχής ABA. Η κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει υπόψη της επίσης και τους στενούς παραδοσιακούς δεσμούς που συνδέουν ε, τους δύο πληθυσμούς. Οι δεσμοί αυτοί θα αποτελέσουν και τη βάση για τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών και μετά το δημοψήφισμα ε, και μετά την 9η Ιουλίου του 2011. Σε ό,τι αφορά την ηθαγένεια τώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι όσοι μεταφερθούν στο βορρά ούτε θα απελαθούν ούτε θα χάσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα σταγένειας που είναι πολύ λεπτό ε, και για το βορρά και για τον νότο, αναμένουμε να πράξει τα δέοντα και η κυβέρνηση για την επίλυση όλων αυτών των ε, ζητημάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή ABA, υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Δεν ε, ξεκίνησε ε, ο πόλεμος για τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Υπάρχουν δεδηλωμένε θέσεις από τις πλευρές. Και φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια ε, συμφωνία. Η έλλειψη ανάπτυξης ε, οφείλε, ε, μάλλον ευθύνεται για πολλά από τα κακά που έχει ζήσει ο σουδανικός ε, πληθυσμό. Ακριβώς η ανάγκη ανάπτυξης ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν και οι προσπάθειες και του Νοτιού Σουδάν. Πρέπει να κινητοποιηθούν πόροι. Έχουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή που απαιτεί βοήθεια. Η διεθνή κοινότητα έχει δεσμευτεί και θα ολοκληρωθούν τα τελευταία βήματα για την βοήθεια αυτή. Επίσης για την παγίωση της ειρήνης και για να υπάρξει ταχεία ανάπτυξη του Νοτιού Σουδάν. Η Ευρώπη θα βοηθήσει και σε ό,τι αφορά το εξωτερικό χρέος. Το χαιρετίζουμε αυτό, αλλά έχουμε τη γενική κατάσταση που αφορά την ειρήνη στην περιοχή και σίγουρα αυτό απαιτεί περισσότερη ε, δέσμευση και ελπίζουμε οι εκκλήσεις αυτές που απευθύνουμε να εισακουστούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ναζάριο τώρα έχει το λόγο. Πέντε λεπτά, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εξοχότητε, ε, αγαπητοί βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω του διοργανωτέ που κάλεσαν την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να ε, δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την πολύ σημαντική ιστορική συγκυρία. Η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν ε, εκφράσει την ικανοποίησή τη με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματο, το οποίο ήταν ειρηνικό και αντικατοπτρίζει την πραγματική δημοκρατική θέληση του λαού του Νοτίου Σουδάν. Οι κάτοικοι του Νοτίου Σουδάν μίλησαν και ξεκάθαρα ψήφισαν υπέρ της θέσπισης ενός ανεξάρτητου κράτους στο Νότο. για την ε, ε, διοργάνωση του αποτελέσματος. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον Ιούλιο του 2011 θα ανακοινωθεί και το ανεξάρτητο κράτος. Εμείς χαιρετίζουμε τη δέσμευση και του Προέδρου Αλμπασίρ και, της, ε, και του Βορρά που είπαν ότι θα αναγνωρίσουν τη βούληση του λαού του Νοτιού Σουδάν και θα συνεργαστούν προς την καθιέρωση και τη συγκρότηση δύο βιώσιμων ε, και ε, αλληλοϊποστηριζόμενων κρατών που θα ζουν ε, ειρηνικά μεταξύ του. επόμενου μήνε, η κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν θα επικεντρώσει την προσοχή τη στην πλήρη εφαρμογή τη ε, CPA, τη ε, Γενική Ειρηνευτική Συμφωνία. Η κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν θα χρησιμοποιήσει τον αναπομένοντα χρόνο τη μεταβατική περίοδου για να συμπήξει στέρεες φιλικές σχέσεις με το Βορρά και θα προσπαθήσει στεναρά να επιληθούν όλα τα εκρεμή ζητήματα το στόματερο δυνατό, ιδίω αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον των σχέσεων βορρά-νότου. Τα ε, δηλαδή, τα σύνορα, το πετρέλαιο και η ασφάλεια, τα βασικά αυτά ζητήματα αλλά πάντοτε με σεβασμό ε, στου όρου ε, τη συμφωνία τη Ειρηνευτικής, η επίλυση αυτών των ζητημάτων δεν είναι προπόθεση για την συγκρότηση του ανεξάρτητου νότιου Σουδανικού κράτου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα ασφαλεία. Αυτά αντιμετωπίστηκαν. Πρέπει να βρεθεί όμω μια μακροπρόθεσμη λύση για την περιοχή ABA το συντομότερο δυνατό. Το Βόρειο και Νότιο Σουδάν έχουν ε, δεσμευτεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου να καταλήξουν σε μια λύση για την περιοχή αυτή. Και εμεί θεωρούμε να, ότι υπάρχουν δύο βιώσιμε λύσει. Η πρώτη είναι να γίνει δημοψήφισμα στην ABA, σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Δεύτερον, με προεδρικό διάταγμα να ε, προσαρτηθεί, να ενταχθεί μάλλον στο Νότο η περιοχή ΑΜΠΑ με βάση ε, και τις αποφάσεις του Εθνικού Διατητικού Δικαστηρίου και του πρωτοκόλου ABA και επίσης με τους διάφορους νομάδες ε, θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και να δώσουμε ε, τους απαραίτητους μηχανισμούς για να υπάρξει επίλυση των προβλημάτων και η πρόσβασή τους ε, στους βοσκότοπους. Η κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν προετοιμάζεται ενεργά για την ίδρυση του νέου κράτους. Θέλει να υπάρξει καλή διακυβέρνηση, δημιουργία υποδομών, θεσμών και επίσης να θεσπιστεί η πλουραλιστική δημοκρατία η, η ειρηνική διεξαγωγή του δημοψηφίσματος είναι ο γνώμονας που δείχνει και τις ικανότητες ε, της κυβέρνησής μας, αλλά και ε, τη σοβαρότητα και την οριμότητα του πληθυσμού μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποια σχέδια για να, γίνει, να θεσπιστεί μια επιτροπή ε, αναθεώρησης συντάγματος. Μετά την ανεξαρτησία η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν θα ε, ζητήσει να γίνει μέλος ε, μεγάλων οργανισμών όπως είναι η ΚΤΑΝΤ, η Αφρικανική Ενότητα, η Κοινοπολιτεία και άλλοι μείζονες χρηματοπιστωτικοί διεθνείς οργανισμοί και σε σημαντικούς μηχανισμούς όπως αυτοί που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η συμμετοχή μας σε αυτούς είναι μία από τις μεγάλες μας προτεραιότητες. και θα θέλαμε και την υποστήριξη για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Η κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο το, Νότιο Σουδάν να ζητήσει να συμπεριθούν και κάποια άλλα θέματα, αλλά πρώτα θα πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το φόρουμ για την ανασυγκρότηση Θέλουμε να υπάρξει υπομονή, γιατί και εμείς θέλουμε πρώτα να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν χαιρετίζει την ε, έγκαιρη δράση από τη εθνική κοινότητα σε ό,τι αφορά το χρέος. Ανεξαρτήτως του πώς ε, θα ε, κατανεμηθεί και ο Βορράς και ο Νότος θα ζητήσουν και θα χρειαστούν διεθνή υποστήριξη για την ανακούφιση του χρέους. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Θα αρχίσουμε με τις ανταλλαγές απόψεων με τους ευρωβουλευτές. Για τρία λεπτά ο καθένας μπορεί να παρέμβει. Να παρέμβει η κυρία Θεοχάρους, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, από τις προσωπικές μου εμπειρίες, τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει κάποιος σε μια επιτροπή ελέγχου ε, ενός δημοψηφίσματος ή εκλογών, ε, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο έργο έχουν επιτελέσει οι συνάδελφοί μας που πήγανε στο Σουδάν σε μια δύσκολη χώρα και θα ήθελα να τους συγχαρώ για αυτό το λόγο. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Μαρία για το μάθημα δημοκρατίας που μας έκανε πριν από λίγο και να εκφράσω την περηφάνεια μου. Νομίζω ότι οφείλουμε να σεβαστούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όχι νομίζω, έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι πρέπει να σεβαστούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και να στηρίξουμε τις χώρες που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος. Να αναπτυχθούν οικονομικά και να αναπτύξουν την δημοκρατία. Δεν γνωρίζω αν η αντίδραση της Ευρώπης θα είναι ενιαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν στηριχτεί η αντίδραση στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η κάθε μια χώρα θα αντιδράσει με τέτοιο τρόπο που στο τέλος θα υπάρξει μια ομοιομορφία στις αντιδράσεις. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, όσο και αν κάποιοι χαμογελάσουν ενδεχομένως και ηρωνικά, ότι και σε αυτό το σώμα και στα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα δημοψήφισμα που έλαβε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο δεν έγινε ποτέ σεβαστό και προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να τιμωρήσουμε τον Κυπριακό λαό για αυτή του την απόφαση. Μην το κάνετε για κανέναν άλλο. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω την Μαρία και την κυρία Ντεκάιζερ. Ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο ότι οι δύο κυρίες ανέλαβαν αυτό το έργο την παρατηρήση των εκλογών και την ηγεσία της αντιπροσωπείας και όπως αναφέρθηκε δεν είναι και εύκολη περιοχή. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι σε μια χώρα που πρακτικά δεν διαθέτει καμία υποδομή, το δημοψήφισμα κατάφερε παρόλα αυτά να λάβει η χώρα με δομημένο τρόπο και το αποτέλεσμα θα είναι πασιφανές όταν θα δημοσιευτεί σήμερα το απόγευμα. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους 60 βοηθούς και παρατηρητές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραβρέθησαν εκεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά και, τους, ε, και τα άτομα τα οποία υποβοήθησαν από το ίδιο το Σουδάν που βοήθησαν και επίσης βοήθησαν και στη φάση καταχώρησης του εκλογικού σώματος το προηγούμενο έτος. Το, τώρα πλέον το δημοψήφισμα θα σημειώσει μια ιστορική στιγμή. Την πρώτη φορά όταν θα αλλάξουν σύνορα στην Αφρική. Τα σύνορα τα οποία όλα προέρχονται πλέον από την αποκεκρατική εποχή και ξέρω ότι ο πρόεδρος του Τσάντ έχει ήδη αναφέρει ότι θα διοργανωθούν εκλογέ στη γειτονική χώρα. Δεν ξέραμε πώ αυτό αποτελεί ένα μήνυμα για περαιτέρω αλλαγέ στα αφρικανικά κράτη. Η πρόκληση του Νοτίου Σουδάν μετά την ανεξαρτησία θα είναι τεράστιε όλε οι προκλήσει που θα αντιμετωπίζει. Πάνω από το 80% του κόσμου είναι αλφάβητοι, 60% ζουν νομαδικά όπως ανέφερα δεν υπάρχουν κανενός είδους υποδομές και οι σχέσεις μεταξύ Νότου και Βορρά θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Τα τελευταία, οι τελευταίες ειδήσει που λαμβάνουμε δεν είναι πολύ θετικές. Υπήρξαν συγκρούσεις με 30 έως 50 ε, νεκρούς στο Βορρά και από το νότιο Σουδάν και στη βόρεια Ουγκάντα ακούμε ότι ενισχύει ο στρατός τα δραστηριότητε του. Επίσης, ένα άλλο ανοιχτό ερώτημα και εδώ νομίζω ότι αυτό αποτελεί πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών στο Νότιο Σουδάν για να δημιουργηθεί ένα είδους κρατικής υπόστασης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε μια πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη και τα υπόλοιπα κράτη, τα γειτονικά κράτη της Αφρικής. Μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί δεν πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να λάβουν χώρα και να γίνουν μέσω των κρατών μελών μεμονωμένα. Όχι. Εδώ αρμόδια είναι η συνολική Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το Σουδάν, για παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Βερονίκη Ντε Κάιζερ και τη Μαρία Ντελτσέπα που ήταν επικεφαλής αυτής της αποστολής, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γνωρίζω αυτές τις ε, δυσκολίες. Ήρθα από τον Ήγηρα, ήμουν επικεφαλής της αποστολής παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν πολλές φορές σε τέτοιες αποστολές παρατήρησης. Εν πάση περιπτώσει δεν θα σας ε, μιλήσω εδώ για το Νίγηρα. Μετά το δεύτερο γύρο θα σας μιλήσω για το Νίγηρα. Θα ήθελα να μιλήσω για την περίπτωση του Σουδάν και ιδιαίτερα σε σχέση με τα σύνορα. Διενεργήθηκε ένα δημοψήφισμα για το ABA. Υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου υπάρχει διχογνωμία, ιδιαίτερα σε σχέση με την περιοχή του Γαλάζιου Νείλου και θα πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους ε, θύλακες και ποιες είναι οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ Βορρά και Νότου. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Τέσσερα σημεία θα ήθελα να θίξω. Καταρχήν η Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία είναι ιδιαίτερα ευφυής και οδήγησε στο δημοψήφισμα. Στάθηκε δυνατόν να τύχει διαπραγμάτευση εξαιτία του μεγάλου ταλέντου των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου της Νορβηγίας και του Ζανγκαράγκ, ο οποίος ε, πέθανε δυστυχώ ε, δύο, ε, λίγες εβδομάδες πριν. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται από το δημοψήφισμα. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές που θα πρέπει να επιληθούν, διότι το Νότιο Σουδάν έχει 2.000 χιλιόμετρα σύνορα με το Βόρειο ο Ελμπεσίρ ήθελε να επιλύσει αυτό το ζήτημα πριν από το δημοψήφισμα και οι εκπρόσωποι του Νότου ήθελαν να επιληθεί εκ των προτέρων. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει επιληθεί. Βεβαίως και στο οικονομικό επίπεδο τα έσοδα από το πετρέλαιο είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει εξωτερικό χρέος το οποίο είναι πολύ μεγάλο και ίσως έχει δημιουργηθεί και ένα προηγούμενο με, βάση αυτό το ε, διχασμό. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να δούμε το νέο κράτος τι ευθύνες φέρει, πώς οριοθετούνται αυτές οι ευθύνες. Μας ενδιαφέρει το πετρέλαιο λοιπόν. Το εξωτερικό χρέος είναι ύψης της σημασίας για να ορίσουμε μια στρατηγική. Άρα το ερώτημά μου ε, στρέφεται προς τους εκπροσώπους του Νοτίου Σουδάν και την Κομισιόν. Τι στοιχεία έχετε για αυτό το νέο κράτος και πώς μπορεί να σταθεί ε, βιώσιμο, να είναι βιώσιμο αυτό το κράτος. Υπάρχει ένα περιθώριο προγραμματισμού Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, γιατί στο Νότιο Σουδάν θέλουμε να ξέρουμε αν είναι λειτουργική η κατάσταση, αν έχουν τα απαραίτητα έσοδα. Χαίρομαι λοιπόν για τον τρόπο διαπραγμάτευσης αυτής της συμφωνίας και εγώ εκπροσώπησα την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 αλλά με απασχολεί το θέμα της βιωσιμότητας αυτού του προγράμματος θα πρέπει να έχουμε αρκετά στοιχεία, χωρίς να μπορούμε να στοιχηματίσουμε, δηλαδή να δούμε όλο αυτό το ευρύ φάσμα μεταξύ του 0 και του 100 και να δούμε πού βρισκόμαστε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ορισμένα στοιχεία ε, εφησυχασμού. Ο κύριος Πάσκου έχει το λόγο. Πέντε λεπτά, όχι παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο άπτεται πολλών πολιτικών πτυχών και στρατηγικών πτυχών. Και δεδομένων των όσων συμβαίνουν στην Βόρεια Αφρική είναι πραγματικά πολύ κρίσιμα τα όσα συμβαίνουν στο Σουδάν. Ελπίζω αυτός, αυτή η ειρηνική διέρεση της χώρας που ανταποκρίνεται στις ε, επιθυμίες του λαού στο νότιο τμήμα να συνεχιστεί και να οδηγήσει σε μια ενίσχυση των θεσμικών ε, αρχών προκειμένου να συνδράμει στην σταθερότητα της όλης περιοχής γιατί η το πρόβλημα θα περιπλακεί περαιτέρω γιατί θα συνδεθεί και με τα υπόλοιπα προβλήματα της περιοχής. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε ίσως τώρα να ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Ναζάρη για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνόρων, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει ήδη με τον Βορρά είναι σημαντικό δηλαδή, συμφωνήσαμε σε σχέση με την χάραξη του 80% των συνόρων της Μεθόριου Βορανότου. Αυτό το οποίο απομένει είναι η περιοχή ABA, ένα τμήμα εκεί και άλλο ένα τμήμα στα βορειοδυτικά ψηλά ε, του Σουδάν, που είναι έτσι αμφιλεγόμενο και αυτό. Η περίοδος που απομένει και για το Βόρειο και για το Νότιο ε, Σουδάν είναι νομίζω αρκετή ώστε οι κυβερνήσεις μας να μπορέσουν να επιλήξουν ε, το ζήτημα των συνόρων. Υπάρχει ισχυρή θέληση των ηγετών και των δύο πλευρών. Και νομίζω ότι αυτός θα είναι και ο λόγος που θα μπορέσουμε ειρηνικά να καταλήξουμε στο θέμα των συνόρων και έτσι να έχουμε εν τέλει αν θέλετε, ειρηνικά ε, και όχι στεγανά σύνορα ε, μεταξύ μας. Σε ό,τι αφορά τον Νότιο Κοτοφάν και τον Γαλάζιο Νείλο, εμείς θεωρούμε ότι οι περιοχές αυτές ε, ανήκουν στο βορρά. Έχουμε ως βάση κληρονομήσει, αν θέλετε, την ανεξαρτησία μας, ε, αλλά είναι στον βορρά αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Ξέρουμε ότι έχουν αγωνιστεί ε, στο, στο πλευρό του SPLA. Έχουν όμως δύο πρωτόκολλα για να επιλύσουν το ζήτημα με την κεντρική κυβέρνηση. Το πρωτόκολλο τους έχει δώσει το δικαίωμα να προβούν σε δημόσια διαβούλευση και είναι σε εξέλιξη στις δύο περιοχές, συγκεκριμένα στο Γαλάζιο γίνεται ήδη και ελπίζουμε και ε, στο νότιο Κοτοφάν να γίνει το ίδιο. Σε ό,τι αφορά την περιοχή τώρα ε, της ABA είναι ε, ένα πρόβλημα μεταξύ των κατοίκων, Οίκονο και Μασυρία συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση όμως του Νοτιού Σουδάν είναι δεσμευμένη στην προσπάθεια να επιληθεί στην, στην εναπομένουσα περίοδο το ζήτημα αυτό της περιοχής ABA. Ε, σας είπα μέχρι το Μάρτιο θέλουμε να έχει επιληθεί το ζήτημα. Ήταν και ένα άλλο ερώτημα που ετέθη. How do we guarantee... Συγκεκριμένα πώς θα εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα του κράτους μας ή τέλος πάντων ποια στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι σήμερα για να μην αποτύχει το κράτος, η προσπάθειά μας. Το πρώτο στοιχείο που έχουμε νομίζω και το οποίο ε, είναι κάτι για το οποίο είμαστε βέβαιοι, είναι η ισχυρή βούληση που έχουμε να μην αποτύχουμε. Υπάρχει ισχυρότατη βούληση έχουμε ισχυρή παράδοση, μεγάλη παράδοση αγώνων στο Νότιο Σουδάν και γι' αυτό και δεν θα αποτύχουμε πιστεύω. parole... Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό εξαχώτησε ο πρέλης του Σουδάν τώρα έχει το λόγο για τρία λεπτά. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Again, I, I, I thank... Θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω τους βουλευτές και όλα τα υπόλοιπα άτομα που συνέβαλαν και όρισαν την ανάγκη περαιτέρω δέσμευσης. Παρατηρήθηκε η ύπαρξη φόβων πριν από το δημοψήφισμα. Αλλά ο Σουδανικός λαός στα νότια της χώρας απέδειξε ότι είχαν τη σοφροσύνη και ότι ήξερε ποιος ήταν ο στόχος τους σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία ακόμα θα πρέπει να λυθούν. Επιβεβαιώνω τη δυνατότητα του Σουδανικού λαού να επιλύσει οτιδήποτε πρόκληση προκύψει. Θα ήθελα να επικεντρωθώ εκ νέου στα θέματα ανάπτυξης. Ο λαός του Σουδάν στο βόρειο τμήμα και στο νότο τμήμα της χώρας είναι αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουν από το στόχο και από το μονοπάτι της ανάπτυξης, την οδό της ανάπτυξης. Σας διαβεβαιώ ότι τα ανεπίλητα ζητήματα δεν πρόκειται να προκαλέσουν πόλεμο στο Σουδάν. Τα δύο μέρη δεν πρόκειται να βρουν διέξοδο στον πόλεμο. Και Πρόκειται για μια πολύ ενημερωμένη απόφαση. Ο λαός του Σουδάν και στα διατμήματα της χώρας θα συνεχίσει στην επιλεγμένη οδό προς την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρόζαλιντ Μάρστιν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, πολύ σύντομα για το θέμα της βιωσιμότητας και ιδίως στο Νότο. Η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν φυσικά έχει τα ενία σε όλο αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος παρέχει 150% εκατομμύρια ε, ως υποστήριξη υπέρ των πιο ευάλωτων πληθυσμών, αλλά θα δούμε και τι αναπτυξιακή βοήθεια θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ε, ιδίως για την δημιουργία υποδομών και θα έχουμε βέβαια σε στενό συντονισμό και με την κυβέρνηση του Σουδάν, αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη και με άλλους αναπτυξιακούς εταίρους. Για τις δημόσιες αυτές διαβουλεύσεις εμείς ε, προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ζήτημα. Με βάση τη γενική ειρηνευτική διαδικασία έχει δοθεί δυνατότητα ε, στους πληθυσμού του Νοτίου Κοντοφάν και στο Γαλάζιο Νείλο να εκφράσουν ε, τη βούλησή τους και θα υπάρξουν στη συνέχεια συστάσεις πρωτοχαρτούμ για να διορθωθούν και ενδεχόμενες αδυναμίες ή ελλείψεις. Είναι μια διαδικασία σωστή. Ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί πριν λήξει μεταβατική περίοδος. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστώ πολύ. Να ξαναδώσω το λόγο στην ε, Μαρία Νεντέτσεβα για πέντε λεπτά. Θα είμαι λίγο πιο σύντομη, δεν θα εξαντλήσω τα πέντε λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάρστιν και τους δύο πρέσβεις πρώτα απ' όλα. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο για ένα ζήτημα που μας ε, ενδιαφέρει σήμερα και μας ε, ανησυχεί και ε, αν ήθελα να κλείσω θα ήθελα να κάνω μια σύνοψη ποια είναι τα τρία μηνύματα τα οποία συγκρατώ εγώ μετά τις παρεμβάσεις των βουλευτών τους οποίους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ειρηνική ατμόσφαιρα, ειρηνικό κλίμα και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Συγκρατώ επίσης ένα μήνυμα που είχαν όλες οι παρεμβάσεις, δηλαδή ότι υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις αλληλένδετες με τις οικονομικές. Και το τρίτο μήνυμα είναι ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο ε, στις ε, Σουδανικές ε, αρχές για να υπάρξει μια ανασυγκρότηση στις δύο χώρες που θα έχουν να κάνουν και κάποιες διαπραγματεύσεις στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ η πρόεδρο. Και εμεί σα ευχαριστούμε για την εξαιρετική σα δουλειά και θα περάσουμε στο σημείο 6. Κυρία Γκρέις δεν έχει έρθει από ό,τι βλέπω. Σα προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 7 τη σημερινή διάταξη και να επανέλθουμε στο 6 εάν και εφόσον έρθει και η κυρία Γκρέις. Συμφωνούμε? Ήρθε η κυρία Γκρέις. Α, Je vous laisse le temps d'arriver, Madame Grèze. Με την ησυχία σας, κυρία Γκρέ, καθίστε.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 S'il Σας παρακαλώ πολύ, συνεχίζουμε. Όσοι δεν θέλετε να παραμείνετε, παρακαλώ να αποχωρήσετε τώρα, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Nous allons Τώρα θα εξετάσουμε το σχέδιο γνώμης της κυρίας Γκρές για την εξωτερική διάσταση της ε, κοινωνικής πολιτικής καθώς και την ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα που αφορά και την εξωτερική πολιτική και την πολιτική πασό. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Άρα αναφερόμαστε στις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσουμε τις κοινωνικές προδιαγραφές στις τρίτες χώρες. Δίνει το λόγο στην κυρία Γκρέζ για 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μας υποβλήθηκε αυτή η γνώμη γιατί η Επιτροπή Απασχόλησης θα ενσωματώσει πολλές από τις προτάσεις που θα υποβάλουμε εδώ και που έχουν σχέση με την ε, απασχόληση. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη προδιαγραφές εργασίας, όχι υπομορφή συστάσεων, αλλά υπομορφή νομικής δέσμευσης, διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε αυτά τα πρότυπα, τα εργασιακά πρότυπα, όταν μιλάμε για μια σταθερή πολιτική και κοινωνική πολιτική σε μια χώρα για να έχουμε καλύτερες εμπορικές σχέσεις. Δηλαδή, όσο πιο δεσμευτικά είναι και δρακόντια είναι τα μέτρα, τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα διασφαλίζουμε για μια χώρα. Ε, Απογοητεύουμε λοιπόν από την έκθεση που έχει υποβληθεί, διότι βρισκόμαστε σε... έχουμε να κάνουμε με μια παρουσίαση όπου υπάρχει μεγάλη προτίμηση στο εμπορικό σκέλος των συμφωνιών, ενώ βλέπουμε ότι οι κοινωνικές διατάξεις δεν τίθενται παρά υπομορφή στόχων, απότερων στόχων. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να θίξω. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να ενσωματώσουμε μια κοινωνική ρήτρα στο σύνολο των εξωτερικών εμπορικών συμφωνιών. Και αυτό αφορά και τις συμφωνίες που έχουν συναυτεί στα πλαίσια του ΠΟΕ. Τρίτον, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες για την θέση σε εφαρμογή αυτών των κοινωνικών προτάσεων διότι πρόκειται για προτάσεις εθελοντικές καθαρά και θα πρέπει να δώσουμε και κίνητρα, αλλά να δούμε ποιες είναι και οι κυρώσεις όταν ε, οι συμφωνίες δεν τηρούνται στα πλαίσια και των διμερών και των πολυμερών συμφωνιών. Τέλος, τέταρτο σημείο, θα ήθελα να μην έχουμε πολλαπλές εξαιρέσεις. Γιατί εδώ μιλώ για τις ελεύθερες ζώνες και τις βιομηχανικές ελεύθερες ζώνες, δηλαδή τις καθαρά εξαγωγικές. Η πέμπτη πρόταση που αφορά τις σχέσεις Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ΠΟΕ οι δύο αυτές προτάσεις σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική αυτών των χωρών και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να προωθούμε παρά τις εμπορικές σχέσεις που προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να μπορεί να προβάλλει ε, ένα εγχείρημα πραγματογνωμοσύνης και σε περίπτωση διαφοράς να υπάρχει μία οδός προσφυγής, κάτι το οποίο δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Το έκτο σημείο αφορά τη λογοδοσία σε περίπτωση παραβίασης. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μία προσέγγιση καθαρά εθελούσια, χωρίς νομική δέσμευση όσον αφορά τις προδιαγραφές εργασίας. Και γι' αυτό ακριβώς συνέταξα μία γνώμη σε σχέση με την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχουν οι βουλευτές και μετά η Κομισιό. Ο κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ. Εδώ μιλώ εξ ονόματος της Πατρίς Τυρολιά που είναι η και θα ήθελα να τονίσω ότι η Κατρίν Γκρέλ ε, τονίζει τη σημασία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και έχεις απόλυτο δίκιο, Κατρίν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσθέσει μια κοινωνική ρήτρα στις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις έτσι ώστε σε επίπεδο ΠΟΕ να μπορέσει να πιέσει για να τηρούνται οι προδιαγραφές Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και στις μας επιχειρήσεις αλλά και ανά τον κόσμο. Η Πατρίς Τυρολία, λοιπόν μου αναφέρει τα εξή πέρα από τα συγχαρητήρια προς εσάς θεωρεί ότι θα πρέπει η κοινωνική διάσταση να γίνει ένας πυλώνας της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μέχρι τώρα η εξωτερική δράση προώθησε τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε την κοινωνική διάσταση της περιφερειακής ολοκλήρωσης που να σταθεί εφαλτήριο στο κοινωνικό αυτό άλμα. Εξάλλου, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι πολυεθνικές να λάβουν υπόψη αυτή τη κοινωνική διάσταση και να τη λάβουν υπόψη σοβαρά όταν μεταβαίνουν στον τρίτο κόσμο. Ε, δηλαδή να, να ληφθούν μέτρα καθαρά δεσμευτικά. Τέλος, τη στιγμή που μιλάμε για κοινοβουλευτική νομιμότητα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, συμμετοχή, να δεχτεί τη συμμετοχή των συνδικάτων και στα πλαίσια του ΠΟΕ και στα πλαίσια των άλλων περιφερειακών διεθνών οργανώσεων και στις περιφερειακές ε, συμφωνίες και τις διμερείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φίζας έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ο Σκιώδης από πλευράς ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι σύμφωνο απόλυτα με την κυρία Γκρές ως προς το έκτο σημείο, δηλαδή την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να οριοθετηθεί αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να εφαρμοστεί το εργατικό δίκαιο αλλά θα πρέπει να υπάρχουν νέοι κανόνες που να εντάσσονται στο εργατικό δίκαιο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα, που βρίσκεται στην αιτιολογική σκέψη της έκθεσης. Είναι η κατάσταση της Κίνας, η παρουσία της Κίνας στην Αφρική. Σας είπα ότι επανήλθα από τον Ήγηρα και εκεί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή η Κίνα αυτή τη στιγμή δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της σε σχέση με το συμβατικό δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως ξέρετε στο Μιονμέι δημιουργήθηκε μία γέφυρα μόνο με Κινέζους εργάτες που βρίσκονται, σε, που βρίσκονται επί τόπου χωρίς να δώσουμε εργασία, να προσφέρουμε εργασία στους κατοίκους του Νίγηρα. Και γίνεται και κοινωνικό dumping κατά των ευρωπαϊκών κανόνων. Γιατί κανείς θα πρέπει να προβάλλει μια διαδικασία διαγωνισμού. Η Κίνα δεν το κάνει αυτό, καθόλου μάλιστα. Οποιοδήποτε ευρωπαϊκό λοιπόν έργο διαρκεί πολύ περισσότερο, γι' αυτό τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να προβάλλουν, να ε, συνάψουν συμβάσεις με την Κίνα, γιατί δεν τηρεί όλες αυτές τις προδιαγραφές και δεσμεύσεις, άρα το έργο τελειώνει πολύ νωρίτερα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τίθενται σε κίνδυνο οι δικέ μας επιχειρήσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες κυρώσεις τη στιγμή που υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα που δεν πληρούν αυτούς τους όρους και πλειοδοτούνται. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να επιβληθεί για να υπάρχουν ίσοι όροι ε, πρόσβαση. Κύρια Θεοχάρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την παρότρινση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της μεταφοράς της ενίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από την σφαίρα του εθελοντικού στην σφαίρα των νομικών υποχρεώσεων. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική διαφοροποίηση που θα δώσει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα γιατί πραγματικά οι λαοί που βρίσκονται σε ανάγκη δεν ε, ξεχωρίζουν αν αυτό που λαμβάνουν ή δεν ρωτάνε ή δεν τους νοιάζει σε τελική ανάλυση αν λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια ή αναπτυξιακή βοήθεια την συγκεκριμένη στιγμή που χρειάζονται την ε, βοήθεια. Γι' αυτό το λόγο, αν σκεφτούμε για παράδειγμα τις φαρμακευτικές εταιρείε και με ποιο τρόπο η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα μπορούσε να μεταφραστεί σε παροχή φαρμάκων για όλους αυτούς που τις, ε, τα χρειάζονται, τότε πράγματι θα έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση για την οποία εργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς. Δύο λεπτά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσ ορισμένες σκέψεις σε σχέση με αυτά που μας είπε. Ζητούμε κοινωνικές ε, δεσμεύσεις που θέλουμε να επιβάλλουμε ανά τον κόσμο. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει αυτό. Σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης υπάρχουν μεγάλα προσκόμματα. Υπάρχει η Κίνα, υπάρχουν οργανώσεις που έχει διαφορετική υπόσταση και ο ΠΟΕ επιβάλλει την τήρηση των ε, κανόνων και δεσμεύσεων κοινωνικού χαρακτήρα, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε επίπεδο διεθνούς ε, γραφείου εργασίας. Δηλαδή δεν πρόκειται για παρόμοια μεγέθη, μάλλον δεν υπάρχουν οι ίδιες δεσμεύσεις σε σχέση με το εμπορικό δίκαιο. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόσχομα. δηλαδή ποιος θα καταβάλει αυτή την προσπάθεια σε επίπεδο διεθνούς οργανισμού εργασίας. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μας πει πώς ε, μπορεί να αναλάβει κάτι τέτοιο, γιατί ως προς εξωτερικές εμπορικές σχέσεις δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Πώς μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο. Πώς θα αποφασίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιος θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρωπαϊ... Εξωτερικής Δράσης έτσι ώστε να εισακουστεί η φωνή της κυρίας Γκρές. Και για να υπάρχει μια αυστηρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η στάση των κρατών μελών, διότι εκείνα δίνουν εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματευτεί τις εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχει λοιπόν μία σειρά εμποδίων που θα πρέπει να αρθούν πριν φτάσουμε σε μία ευρωπαϊκή κοινή θέση. Μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερος κοινωνικός χαρακτήρας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά μέχρι που, ποιο σημείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει μάχη με τους άλλους διαπραγματευτές πώς θα δείξει την πυγμή της. Ο κύριος Μαρτίνες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως φαίνεται λογικό και σε σχέση και με αυτά που είπε και ο συντονιστής μου, ο κύριος Μπέρμαν, νομίζω ότι συμφωνούμε και στις τοποθετήσεις και στις προθέσεις και στην βούληση να σημειωθεί πρόοδος. Αυτό άλλωστε νομίζω ότι διατρέχει όλες τις συστάσεις της φίλης ε, Γκρές στην έκθεσή της. Τώρα, νομίζω ότι θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση γιατί θέλω να σας πω το εξής. Ε, στις χώρες αυτές, οι χώρες αυτές έχουν υπογράψει τη συμφωνία. Συνήθως μιλάμε μακριά από το μικρόφωνο ο μιλητής. Εάν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει συνέπεια από τις χώρες οι οποίες προσυπέγραψαν συμβάσεις ε, της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πρέπει να τηρούνται. Άρα το θέμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι σημαντικό. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θέλω να αναφέρω. Εγώ πάντοτε ε, βρίσκομαι σε αμήχανη θέση γιατί η κοινωνική ρήτρα όπως η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ρήτρε οι οποίες φαίνεται ότι τις έχουμε συμπεριλάβει στις ε, συμβάσεις ε, έτσι για να έχουμε ε, ήσυχη τη συνείδησή μας. Έχουμε λοιπόν ρήτρα ανθρώπινων δικαιωμάτων με χώρα που θα μπορούσαμε... Έχουμε χώρα, ρήτρα αυτή με το Ισραήλ, παραδείγματο χάρη, μια χώρα η οποία συνέχεια παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τα κατεχόμενα, το, τα εδάφη, τον Παλαιστινιακό λαό. Λοιπόν, όχι επί σειρά ετών ε, που είχαμε σε ισχύ αυτή τη ρήτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί, αλλά δεν έχει υπάρξει ε, κανένα αποτέλεσμα. Ούτε καν δεν έχει συγκροτηθεί το όρο το οποίο θα ε, μελετούσε ενδεχομένω κάποιε κυρώσει όταν έχουμε αυτή τη συστηματική συμπεριφορά σε σχέση με τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με μια χώρα σημαντική φίλη κτλ. Που όμω φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο καμία άλλη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε δεν έχει άλλη αξία αποτελικά να είναι μια ε, διακήρυξη. Καλό είναι αυτό, εντάξει, να κάνουμε διακήρυξεις ε, καλών προθέσεων κτλ. Αλλά μην ε, κοροϊδευόμαστε. Μην αυταπατώμεθα νομίζοντας ότι αν εισαγάγουμε κάποιες ρήτρε θα αλλάξουν τα πράγματα. Άλλο είναι η δεύτερη οργάνωση εργασία, γιατί αυτό το οποίο θα μπορούσε να απαιτήσουμε είναι χώρε που έχουν προσφογράψει τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να τις εφαρμόζουν τα συμβάσεις αυτές. Αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Κύριος ή κυρία Τάμας Βάρνης, δεν ξέρω, λέει η πρόεδρος. Κυρία, περί κυρίας πρόκειται, μάλιστα. Κριστίν Σράιμπερ λέγομαι, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόλησης. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας υπογραμμίσω πόσο εκτιμούμε το θέμα ότι το Κοινοβούλιο μιλάει για το θέμα αυτό της εξωτερικής πολιτικής στο, στην γνωμοδότησή του και το γεγονός ότι η Επιτροπή σας ε, καταρτίζει γνωμοδότηση, ο συνεχής διάλογος στους τομείς αυτούς είναι, θεωρώ, και σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο ουσιώδης σημασία. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που έθιξε και η συγγήτρια, αλλά και κάποιοι βουλευτές για τις ε, εμπορικές συμφωνίες. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αξιόπιστη, την ε, έντιμη εργασία μέσω των εμπορικών πολιτικών, μέσω των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και των συμφωνιών επένδυσης. Πρόσφατα αντιπραγματευτήκαμε τέτοιε ε, ε, συμφωνίες ελεύθερης ζώνης εμπορίου και ζητήσαμε να δεσμευτούν και όλες οι πλευρές προς τα υψηλά πρότυπα εργατικά και σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών και στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να επικυρώσουν τη Σύμβαση για τα Κριτήρια Εργασίας της Διεθνής Οργάνωσης, Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας που ισχύουν σήμερα. Άρα είναι πολύ εντατική η συνεργασία μας και με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, όπως ανέφεραν και οι βουλευτές. Για τον μηχανισμό εφαρμογής τώρα, η ε, Κομισιόν βασίζεται στην συνεχή δέσμευση και διάλογο με τα εμπλεκόμενα μέρη. Με έναν μηχανισμό αξιολόγησης και ελεύθερης συμμετοχής είναι πιο πιθανή η επιτυχία παρά με έναν μηχανισμό κυρώσεων. Ωστόσο, ασφαλώς η Κομισιόν είναι διτεθειμένη να συζητήσει και τέτοια θέματα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προτύπων των περιβαλλοντικών και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το CSR που διάφοροι βουλευτές ανέφεραν. Η ανακοίνωση που εγκρίθηκε το 2006 διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια εθελούσια ε, συμφωνία που καλεί τις επιχειρήσεις να είναι πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνε, αλλά έχουν αλλάξει και έχουν εξελιχθεί τα πράγματα έκτοτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξελιχθεί η έννοια της εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Δεν θα απέκλεια συμπληρωματικά μηχανισμούς και συμπληρωματικές δράσεις πέρα από το βασικό μηχανισμό. Και Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκρέσ για τρία λεπτά για να καταλήξει με τη συζήτηση. Παρακαλώ. Έχετε ένα ερώτημα. Εκτάκτως επειδή είστε εσείς θα σας δώσω το λόγο, κύριε Μπέρμαν. Νομίζω ότι καταργήθηκαν ε, τα προνόμια μετά το 89. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε σχέση με το monitoring, κάποια δεσμευτικά μέτρα, δεν κατάλαβα καλά τι εννοούσατε και θα ήθελα να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί και εγώ, εδώ και δύο χρόνια, αγωνίζομαι για να γίνουν από πλευρά τη Επιτροπή αυτό που θεωρώ πολύ απαραίτητο, δηλαδή να καταπολεμηθεί η παιδική εργασία σε μια χώρα ε, υπό ανάπτυξη και αυτό μεταξύ άλλων μέσω ενό δεσμευτικού μέτρου που θα ήταν πολύ απλά η καθίδρυση ε, μιας τηλεφωνικής γραμμής, hotline, που θα είναι ανοιχτή προς όλες τις οργανώσεις και προς όλα τα άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και αλλού, που θα μπορούν ε, να δηλώνουν να αναφέρουν τέτοια κρούσματα. Όταν υπάρχει δηλαδή κατάχρηση μιας ε, κατάστασης, ε, όταν δεν υπάρχουν ε, καθόλου είτε αρκετά τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως στην ακτή του ελεφαντοστού, που η συλλογή του κακάου γίνεται στο μεγαλύτερο βαθμό από παιδιά. Και οι σοκολάτες αυτές έρχονται στην Ευρώπη και δεν λέει κουβέντα κανένας και δεν κάνει τίποτε κανένας. Ίσως για την απασχόληση στην Ευρώπη να είναι καλό αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ κακό για την ανάπτυξη αυτών των αναπτυσσόμενων χωρών. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να είμαστε πολύ πιο δεσμευτικοί, γιατί πρέπει να αφυπνιστεί η κοινή γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα και πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική παρακολούθηση, αυτό το monitoring που είπατε, μέσω και αυτή τη γραμμή τη τηλεφωνική. Θα ήθελα να δώσετε λεπτομέρειε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, λοιπόν, πρόεδρο, έχουμε 10 λεπτά καθυστέρηση. Ε, θα δώσω ένα λεπτό στην Κομισιόν <clears throat> για να απαντήσει. Και βέβαια μπορείτε και διμερό ενδεχομένω στη συνέχεια να το δείτε. Έχετε ένα λεπτό. Θα απαντήσω πολύ γρήγορα, λέει η Κομισιόν, και ίσω μετά θα μπορούσαμε διμερό να τα πούμε για περισσότερε λεπτομέρειε. Έχουμε το επίσημο πλαίσιο πρώτα απ' όλα. Αν έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίο αυτομάτω βασίζεται σε κάποιε ποινέ ε, ή σε αναστολή ε, των ε, κερδών κτλ. στο πλαίσιο τη Συμφωνία Εμπορίου ή από την άλλη προτιμούμε ένα πιο ευέλικτο μηχανισμό με κάποιες ανεξάρτητες επισκοπήσεις, ε, αναθεωρήσεις, ε, με τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων, γιατί νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα μόχλευσης με αυτόν τον τρόπο παρά μόνο αν έχουμε έναν μηχανισμό ή όλα ή τίποτα. Αυτό που λέτε βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πολλές δυνατότητες για να ειδοποιήσουμε, να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου αν υπάρχουν ε, τέτοια κρούσματα παιδικής εργασίας κτλ. Μπορούμε να ασκήσουμε τις πιέσεις μας και τις δυνατότητες μόχλευσης που έχουμε με τις ε, διάφορες χώρες αλλά θα έλεγα να το συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα, και με τους συναδέλφους από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο, που είναι η καθήλυνα αρμόδια γενική διεύθυνση. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκρέσ με δύο-τρία λεπτά έχει τη διάθεσή σα. Εντάχει, σα ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια που ακούστηκαν, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σημασία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και την ε, κοινωνική πολιτική που θα γίνει ένας από τους πυλώνες της ε, εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης. Το θέμα της Κίνας και της Ασίας πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Το να χρησιμοποιούμε το παράδειγμα της Κίνας και της Ασίας για να μην κινηθούμε προς δεσμετυπτικά μέτρα, αυτό σημαίνει ότι καταδικάζουμε τον εαυτό μας κάθε φορά τη στιγμή που φτάνει μια νέα χώρα με χειρότερες κοινωνικές συνθήκες, δηλαδή ο πύχης κατεβαίνει ολοένα και προς τα κάτω σε σχέση με τον απότερο στόχο μας, για να υπάρχει δηλαδή μια καλύτερη αναπτυξιακή πορεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πολιτική σταθερότητα, αλλά να υπάρχει και καλύτερη κατάρτιση, περισσότερες αρμοδιότητες και μία ενδογενή ανάπτυξη των χωρών αυτών. Αυτά ήθελα να σας πω με λίγα λόγια. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών ορίζεται για τις 10, στις 10 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 22 Μαρτίου στην ε, συνεδρίασή μας. Τώρα θα γίνει η συζήτηση για τη νέα εμπορική, ε, ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Όπως ξέρετε, στόχος είναι να ενισχύσουμε το εμπόριο υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή λοιπόν το εμπόριο είναι ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την αναπτυξιακή πορεία, ζητήσαμε τη σύνταξη μιας έκθεσης έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η συνοχή από την ίντα. Η κυρία ε, Μπρίζιτ ε, Σνίμπερ Ζάστρα με έχει το λόγο για να μας ε, μιλήσει για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής συνοχής. Ήταν αδύνατον στην γνωμοδότηση αυτή, λόγω χωρικών περιορισμών, να αναφερθούν όλα τα στοιχεία. Γι' αυτό, λοιπόν, και ευγνωμονώ ιδιαίτερα για ενδεχόμενες, τις ενδεχόμενες ε, προσθήκες σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της εμπορικής πολιτικής της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ό,τι αφορά την πτυχή, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική το 2020, θα θυμάστε ότι το 16 Μαρτίου του προηγούμενου έτους ο ε, Επίτροπος Δεχούχτ είχε πει ότι μακροπρόθεσμο το εμπόριο θα πρέπει να συμβάλλει προκειμένου όλοι οι κάτοικοι της γης να, να βελτιώσουν την ύπαρξή τους και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνεται εμφανώς αυτή η πρόθεση. Μία ρητή αναφορά στην πολιτική συνοχής είναι απαραίτητη και αυτό νομίζω ότι διευκρινίζεται στους παραγράφους 1 και 2 επειδή για παράδειγμα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό του εμπορίου δεν αποτέλεσε αυτό θέμα πυρήνα και βασικά επικεντρωνόμαστε στα θέματα των ευρωπαϊκών εταιριών και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στη διεθνή αγορά. Και επίσης προστίθονται μέτρα τα οποία σκοπό έχουν να εγγυηθούν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες και σε δημόσιους διαγωνισμούς για προμήθειες. Η βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται μεν στην ανακοίνωση, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τα θέματα οικολογίας. Οι λοιπές πτυχές της βιώσιμης και αποδοτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνουν για παράδειγμα οικονομικά, κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα ε, ουσιαστικά δεν αναφέρονται, δεν υπογραμμίζονται στην ε, ανακοίνηση και επίσης αναφέρεται το policy space ε, στην ανακοίνωση, ένα περιθώριο ελιγμού που χρειάζονται οι χώρες για να καταπολεμήσουν την ένδια, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει ο νότος, ε, το νότιο ημισφαίριο να οικοδομήσει σωστές αγορές. Ένα άλλο θέμα θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως η πρόσβαση στην ε, η ιατρική υποστήριξη πρωτοβουλειών ιδιωτικών, το οποίο είναι φυσικά ευκταίο. Πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα γενώσιμα φάρμακα και τα ίδια ισχύουν και για τον τομέα, για τον κλάδο των πρώτων ήλων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρούμε τις επιχειρήσεις αυτές όχι ως αντιπάλους αλλά ως εταίρους. Υπάρχει η θέληση όπως φαίνεται από πρωτοβουλίες, όπως ε, η χάρτα εθνικών, ε, φυσικών πόρων και άλλες, γιατί γνωρίζετε ότι οι σημερινές ε, αναπτυσσόμενες, μάλλον οι σημερινές αγορές που χαρακτηρίζονται από φτώχεια είναι οι αυριανές αναπτυσσόμενες αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν ζητάει κανένα το λόγο. ο κύριος Μαρτίνες για δύο λεπτά. Θα ήθελα να πω ότι γενικά συμφωνώ με τις υποδείξεις της συναδέλφου. Έχει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα υπογραμμίζει. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα ως προς το σημείο 4 των προτάσεών της, η πρώτη πρόταση λέει ότι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει ε, ορισμένα ε, προσκόμματα ή εμπόδια τα οποία δεν είναι τελωνιακού ή δασμολογικού χαρακτήρα. Όταν μιλάμε για μη δασμολογικού χαρακτήρα μπορεί κανείς να σκεφτεί τις επιδοτήσεις στις χώρες μας και στη συνέχεια αναφέρεται ότι ότι ε, σε σχέση με τις ε, δασμολογικές επιβαρύνσεις, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, από τη μία μιλάμε για την ε, μείωση μη δασμολογικών εμποδίων και στη συνέχεια μιλά για έναν τύπο επιβαρύνσεων που είναι καθαρά δασμολογικού χαρακτήρα. Δηλαδή, το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε θα ήταν να παραμείνουμε στο να αρκεστούμε στη μείωση μη δασμολογικών επιβαρύνσεων. Νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα περίπλοκο για τις περισσότερες χώρες. Αλλά αν ζητάμε μείωση μη δασμολογικών εμποδίων και στη συνέχεια μιλάμε για επιβαρύνσεις σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος είναι σαν να έρουμε το πρώτο τμήμα της πρότασης. Εν πάση περιπτώσει η πρόταση είναι άκρος ενδιαφέρουσα και θα θέλαμε να δούμε κατά πόσο το Διεθνές Γραφείο Εργασίας θα λάβει υπόψη τις υποδείξεις Η κυρία Γκρέσ για δύο λεπτά ή ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ εντάχει. Η συνάδελφος ήταν σκιώδης η συνάδελφος που ήταν σκιώδης ε, δεν είναι παρούσα. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω τρία σημεία. Καταρχήν, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συνοχή δυνάμει του άρθρου 208 το να λάβουμε υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την προστασία του περιβάλλοντος και την εξόριξη πρώτων υλών που να σέβεται το περιβάλλον. Θα ήθελα όμως να υποβάλω με ένα σχόλιο και να πω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες αηφόρου ανάπτυξης ή βιώσιμης ανάπτυξης που δεν ορίζονται επί του παρόντος. Δεύτερον, στο κείμενο δεν υπάρχουν επιφυλάξεις σε σχέση με το, με το ΠΟΕ, με τον ΠΟΕ, δηλαδή ως προς τα, ε, φυτο, τα ε, προϊόντα connaissance du de précaution. Με τα φυτοφαρμακευτικά προϊόντα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό το κείμενο μιλά για την απελευθέρωση των υπηρεσιών Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ισχύει κάτι τέτοιο στις πλέον αναπτυγμένες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι πολιτικές μας είναι συνεπείς. Μιλάμε για μια στρατηγική που βασίζεται σε ένα πρότυπο, εξαγωγικό πρότυπο καθαρά, χωρίς να λάβουμε υπόψη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Και θα ήθελα να πω ότι μια εμπορική πολιτική δεν μπορεί να κινηθεί κατά του περιβάλλοντος και των κοινωνικών προδιαγραφών. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Βαν Βίνσεν για ένα λεπτό. Καλημέρα. Είμαι ο επικεφαλής, ο αναπληρωτής διευθυντής ε, για τις πολιτικές συντονισμού. Θα σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η Επιτροπή ευχαριστεί την Επιτροπή ε, Ανάπτυξης για το ενδιαφέρον που καταδεικνύει και όπως τονίζεται στην ομαδότηση, όντως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η πολιτική εμπορική είναι συνεκτική και συνεπής σε ό,τι αφορά και τις άλλες ε, πολιτικές και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η Επιτροπή σας να εξετάζει τα θέματα αυτά και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή η ίδια η ανακοίνωση τονίζει το θέμα της συμπερίληψης της εμπορικής πολιτικής. Άρα οι πτυχές της ανάπτυξης έχουν ληφθεί υπόψη και μάλιστα με τον αυτό τρόπο. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση όντω συνάδει με το όλο πνεύμα της ε, ανακοίνωσης. Μπορεί να έχετε διαπιστώσει ότι ναι, μεν δεν τονίζονται στην ανακοίνωση ε, τα θέματα της ανάπτυξης τα έχουμε σημειώσει γιατί όπως θα ξέρετε μέχρι τα τέλη του έτου σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε ανακοίνωση ειδικά για θέματα περιβάλλοντος. Άρα εκεί θα αναπτύξουμε περαιτέρω τις ιδέες που επιγραμματικά αναφέρονται στην τρέχουσα ανακοίνωση και θα εξετάσουμε ζητήματα όπως η προνομιακή μεταχείριση, η διαφορετική μεταχείριση, ε, η αρρωγή, η εμπορική και το καθεξής. Σε ό,τι αφορά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης έγινε μια συζήτηση στην οποία δεν θέλω να επανέλθω, αλλά να υπογραμμίσω το εξής. Το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης του Φόρουμ, μια σημαντική συμφωνία με τις χώρες της Κραϊβικής, μια σημαντική εμπορική αλλά και αναπτυξιακή συμφωνία Σας έδωσα ένα λεπτό και έχετε ξεπεράσει τα δύο. Α, δεν το είχα καταλάβει. Θα ολοκληρώσω λοιπόν ε, με αυτήν την ε, αναφορά μου στη συμφωνία με το Κάρι Φόρουμ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε το λόγο για να ολοκληρώσετε, συνάδελφε, ή όχι. Δεν θέλω να πω τίποτα κλείνοντα, γιατί θα το συζητήσουμε. Okay. Okay. Euh, Ωραία. Επομένως, α, ξέχασα να σας πω, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 14 Φεβρουαρίου, θα ψηφίσουμε την 3η Μαρτίου, στις 3 Μαρτίου στη συνεδρίασή μας. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 8 της μερίσιας διάταξης. Πώς θα αυξηθεί λοιπόν η αποτελεσματικότητα της αθλητικής πολιτικής, εισηγητής ο κύριος Κατσμάρικ. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων, λοιπόν. Περιμένουμε μια, έκθεση, μια ανακοίνωση από την Κομισιόν, μια πράσινη βίβλο συγκεκριμένα Θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις ε, για την Πράσινη Βήλο. Θα συζητηθούν και στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ανάπτυξης 22 Φεβρουαρίου και η δημοσίευση της ανακοίνωσης Επιτροπής ε, που θα επακολουθήσει ανακοινώθηκε για τον Ιούλιο. δεν είναι διαθέσιμο παρά μόνο στα αγγλικά δυστυχώς αυτό το έγγραφο. Όταν θα είναι έτοιμες μεταφράσεις θα τις λάβετε. Και η ΝΤΕΒ έχει ζητήσει να διεξαχθεί μια μελέτη από εμπειρογνώμονες, μελέτη η οποία είναι σήμερα διαθέσιμη για όλους τους βουλευτές. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κατσμάρεκ τώρα, που θα παρακαλέσω να είναι και σύντομος. Zielona Księga jest e, ambitna, już sam είναι πολύ φιλόδοξη η έκθεση αυτή που μιλάει για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας που δείχνει και την ε, μεγάλη φιλοδοξία που πρέπει και να την υποστηρίξουμε. Νομίζω ότι η πράσινη βίβλος είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας για να δοθεί νέα πνοή στη συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή πολιτική, πώς να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις. Ωστόσο η πράσινη αυτή βίβλος νομίζω ότι επιβεβαιώνει και την εγκυρότητα των βασικών μας αξώνων δράσης. Δηλαδή, προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι η ανάπτυξη και η αναπτυξιακή στόχη. Και στηρίζουμε όλες ε, τις ε, δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια. Η πράσινη βίβλωση επίσης προτείνει να ε, επικεντρωθούμε σε κάποιες νέες πτυχές που έχουν σχέση με την αλλαγή του κλίματος και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη γεωργία. Για την εκπόνηση αυτού του εγγράφου εργασίας, εγώ θα επικεντρωθώ σε ορισμένες πτυχές που θεωρώ ότι είναι σημαντικές, και για τις οποίες νομίζω χρήζουν είτε διευκρινήσεις είτε υπάρχουν κάποιες ε, ασάφειες ό,τι αφορά τον ορισμό ή την ορολογία εν γέννη. Πρώτον, σχεδιασμός ή χάραξη μιας άκρος αποτελεσματικής πολιτικής, το άκρος υπογραμμισμένο. Δεύτερον, σχεδιασμός μιας οικονομικής ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει την κοινωνική ανάπτυξη. Πρώτη πτυχή λοιπόν, άκρος αποτελεσματική πολιτική. Φυσικά και θέλουμε όλες οι πολιτικές της Ένωσης να είναι άκρος αποτελεσματικές. Στη διατύπωση αυτή νομίζω ότι υπάρχει έτσι και ένα ρητορικό στοιχείο αν θέλετε Κάποιες φορές όταν χρησιμοποιούμε, λέμε στη χώρα μου, την Πολωνία, τόσο πολύ βαρύγδουπες ε, εκφράσεις, ε, στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα. Ε, άρα δεν μας ενδιαφέρει εδώ τόσο η ρητορική, αλλά η πρακτική εφαρμογή. Γνωρίζουμε το εύρος της φτώχειας στον κόσμο και αν συγκρίνουμε το εύρος της στόχιας με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι πραγματικά ε, εύκολο να συνειδητοποιήσει κανείς πόσο λίγοι πόροι υπάρχουν για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και διάκρος αποτελεσματικά αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ορισμένες συγκεκριμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, επί παραδείγματι καλύτερο συντονισμό, τη θέμενη αξία, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ή μόχλευση και επίσης καλύτερη αξιολόγηση. Όλες αυτές οι δράσεις ε, είναι καλές, ε, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην ε, δώσουμε απόλυτο χαρακτήρα σε αυτές τις αρχές, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα επικεντρωθούμε μόνο στις χώρες που Εντό εισαγωγικών είναι εύκολο ε, να μας δώσουν όλους αυτούς τους δείκτε. Οπότε μπορούμε να πούμε να ορίστε είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε όμως και χώρες πολύ φτωχέ, τις πλέον φτωχέ χώρες, που δεν είναι τόσο εύκολο να επιτύχουμε τους δείκτε αυτούς. Παραδείγματο χάρη, το Νότιο Σουδάν, για το οποίο μιλήσαμε μόλι πριν. Είδα ότι υπάρχουν ε, καταγγελίες ε, και παράπονα από αφρικανικές οργανώσεις για, το, για τη δύσκολη πρόσβαση. Διότι το Νότιο Σουδάν δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ε, αργό, την δική ορολογία που χρησιμοποιείται στις αιτήσει κτλ. Όμως οι πιο πλούσιες χώρες είναι πιο αποτελεσματικές από την άλλη σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα έγγραφα, τι αιτήσει, τα έντυπα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Επομένως δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για αυτές τις χώρες. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό σε σχέση πάντα με την αποτελεσματικότητα, την άκρα αποτελεσματικότητα, είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις διάφορες προτάσεις της στο δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους ε, στη συνάντηση ψηλού επίπεδου. Η Πολωνική Προεδρία επίσης θα ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τη στήριξη του Συμβουλίου, τουλάχιστον επί Πολωνικής Προεδρίας για αυτό το θέμα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θέλω να αναφέρω και το οποίο το έχουμε συζητήσει είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης φυσικά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό και τη μεγαλύτερη ομοιογένεια της πολιτικής, αλλά αυτό είναι ακόμη δυνητικό. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε αν πράγματι ο συντονισμός θα βελτιωθεί και αν η πολιτική αυτή θα γίνει πιο αποτελεσματική. Μια άλλη πτυχή είναι η ανάπτυξη για όλους, inclusive development. Πρόκειται για μία πρόταση η οποία αποσκοπεί στην προώθηση μιας βιώσιμης αηφόρου ανάπτυξης που θα λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι δύσκολο να πούμε σε τι ακριβώς θα συνίσταται αυτή η πολιτική που θα αποσκοπεί στην πρόθεση αυτή του είδους της ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στον ενεργό πληθυσμό ή στον βιοδραστήριο πληθυσμό που έχει ευκολία πρόσβαση και μπορεί να χρησιμοποιήσει τους καρπούς της ανάπτυξης να τους αξιοποιήσει καλύτερα, πρέπει να ε, σκεφτούμε τους πλέον ενδύσεις, τους πλέον φτωχούς που και αυτοί θα πρέπει να ωφεληθούν. Επομένως η ένταξη, η συμπερίληψη είναι μια τεράστια πρόκληση γιατί μιλάμε για την ένταξη στην αγορά εργασίας, μιλάμε για την οικοδόμηση ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας, φορολογικό σύστημα για όλους κτλ. Είναι δύσκολα, απαιτητικά όλα αυτά τα καθήκοντα. Και βέβαια υπάρχει θετική πτυχή και όψη της ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δύο είναι οι σημαντικότερες πτυχές πάντοτε. Η παιδεία και η υγεία. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ένταξη αν δεν υπάρχει πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία. Και για να ολοκληρώσω δύο λόγια ακόμη. Αυτό που έλεγα στην αρχή ουσιαστικά θέλω να επαναλάβω. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε παλαιότερα. Δεν μπορούμε ε, να ξεχάσουμε αφήνοντα κατά μέρο δηλαδή τα παλιά προβλήματα και τις παλιές δεσμεύσεις, να ασχοληθούμε με νέα προβλήματα και νέες δεσμεύσεις. Επίσης, κάποιες διορθώσεις, οι αλλαγέ στην αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι κάτι μονόπλευρο, γιατί εδώ μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ τριών θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Θα ήταν κακό να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα μόνο μερό. Επίσης, η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να είναι εύληπτη, να είναι κατανοητή για τον απλό πολίτη γιατί μόνο έτσι θα στηρίξουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτή την πολιτική. Η γλώσσα με την οποία περιγράφουμε αυτή την πολιτική είναι δύσκολη. Δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος. Και αυτό που μετράει είναι η αποδοχή των πολιτικών μας από τους πολίτες. Πρέπει οι πολίτες μας να γνωρίζουν για ποιο λόγο προσφέρουμε αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει και η εκπαιδευτική πτυχή να έχει την απαραίτητη προσοχή. Και περιμένω βέβαια τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε σε ένα δεκάλεπτο, γι' αυτό θα δώσω λόγο στην κυρία Σνίπερ για ένα λεπτό. Ένα μισή λεπτό. Ζήτησε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί είναι πραγματικά πολύ καλά καταρτισμένη η έκθεση. Και επίσης να τον ευχαριστήσω που θέτει το θέμα της πολιτικής συνοχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το EID. Γιατί είναι σωστή η υπόδειξη σε ό,τι αφορά την πτυχή της ανάπτυξη της ανάπτυξης, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα για την ανάπτυξη με την πτυχή, αν θέλετε, την πολιτισμική, την πολιτική, την ε, κοινωνική σε ό,τι αφορά θέματα αποδοτικότητας. Επίσης, είναι σημαντική η υπόδειξη ότι δεν ε, πρόκειται μόνο αποκλειστικά δηλαδή για θέματα ανάπτυξης, όπως είπατε, αλλά το θέμα είναι η ποιοτική ανάπτυξη σε ό,τι αφορά και την κατανομή. Τη σωστή. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ και πάλι είναι πραγματικά πολύ καλό το έγγραφό σας. Ο κύριο Μπέρμαν για μισή λεπτό. Θα προσπαθήσω να αρκεστώ σε αυτό το χρόνο. Έχετε και το σφυράκι σας σε περίπτωση ανάγκης. Σας ευχαριστούμε Φιλίπ για την ε, πολύ καλή δουλειά στο οποίο περιλαμβάνονται, στο έγγραφο σου περιλαμβάνονται τα πιο, βασικά, τα πιο πολλά βασικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά όμως τη συνοχή, σε ό,τι αφορά την ε, συνοχή της πολιτικής, συνήθως μιλάμε για την αναπτυξιακή πολιτική και σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο και την ε, πολιτική, την αγροτική. Σπάνια μιλάμε για πολιτική συνοχή σε ό,τι αφορά την ε, πτυχή της εξωτερικής πολιτικής. για τα τεράστια έργα ανάπτυξης στα οποία συμμετέχουν ε, πάρα πολλοί άνθρωποι και συμμετέχουν και συνεργάζονται με τους ε, ηγέτες ε, άλλων χωρών ενώ οι ηγέτες αυτοί τελικά καταλήγουν να στέλνουν χρήματα στη Γενέβη σε διάφορες τράπεζες και συνεχίζουν να υπάρχουν ανισότητες. Αυτή η συνοχή που χρειάζεται προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας, της αναψυξιακούς, θα πρέπει να τονίζεται πιο συχνά, γιατί στα κράτη μας ε, είναι όλο πιο έντονη η κριτική που ασκείται κατά της αναπτυξιακής βοήθειας και υπάρξει επίσης μεγάλη απογοήτευση γιατί πολιτική ή εξωτερική μας δεν μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει σε επίπεδο αναπτυξιακή πολιτική. Και το συζητήσαμε αυτό και με τον Επιτροπό Πίμπαλξ και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Εν μέρη και χάρη στο εγγραφό σου, Φίλιπ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Μαρτίνε για 1,5 λεπτό, λέει πρόεδρο. Ευχαριστώ. Εγώ δέχομαι απόλυτα αυτά που είπε ο κύριος ε, Μπέρμαν σε σχέση με τη συνοχή και θα ήθελα να συγχαρώ τον Φιλίπ γιατί θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε κατά τον ε, μεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Μιλάμε για συνοχή αξιών, δηλαδή μία στιγμή με τη συνθήκη της Λισαβόνας, εισαγάγουμε την αρχή αλληλεγγύης μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πιστεύω ότι αυτή, αυτό δεν μπορεί να γίνει για λόγους καθαρά εσωτερικής χρήσης, δηλαδή τη στιγμή που προβάλλουμε αυτό το έμβλημα προς τα έξω. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενταχθεί και αυτό στην ε, έκθεση. Υπάρχει μία πρόταση, Φιλίπ, που θα ήθελα να αλλάξει. Είναι η τελευταία σελίδα 3, όπου λέει ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την αρχή της αλληλεγγύης, ακόμα και μία, κατά μία περίοδο κρίσης. Θα πρέπει να πούμε ότι όμως ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την αρχή της αλληλεγγύης ειδικά σε καιρούς κρίσης. Γιατί τότε είναι πιο δύσκολη η αλληλεγγύη αλλά και ολοένα και πιο αναγκαία. Επίσης, στο έγγραφο αυτό, το οποίο διάβασα διαγώνια, δεν είδα να γίνεται λόγος για το φόρο διεθνών συναλλαγών, επί των διεθνών συναλλαγών, ως μηχανισμό για τη δημιουργία εσόδων μέσα στα πλαίσια εξέβρεσης πόρων για την συνεργασία προς την ανάπτυξη. Αυτό θα ήταν απόλυτα αναγκαίο, διότι όλοι έχουμε δεσμευτεί ως προς αυτό το μηχανισμό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους μας έτσι ώστε η ανάπτυξη να γίνει και να γίνει ακόμη πιο γρήγορα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστώ και τους συνάδελφους. Κύριος Ντόιζερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να, συγχαρώ, να σα συγχαρώ, μάλλον, Πρόεδρε, γιατί ακολουθείτε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα. Κατά δεύτερον, επί της αρχής. Είναι καλό το γεγονός ότι μας υποβάλλει η Πράσινη Βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έκθεση του συναδέλφου είναι πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ατζέντα της αποδοτικότητας της βοήθειας και να πω ότι όλοι θέλουμε πιο μεγαλύτερη αποδοτικότητα και η διακήρυξη του Παρισίου των Παρισίων ήταν ένα πρώτο βήμα πριν από πέντε χρόνια. Αυτά που αποφασίστηκαν επίσης εγώ ελπίζω να υπάρξουν εξελίξεις και πρόοδος αν συνεχίσουμε τον ε, δομημένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ψηφιστούν τα σχετικά προγράμματα το Μάιο υπό την Αγγλική Προεδρία. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία. Αφενός, όταν επισκεπτόμαστε χώρες ανάπτυξης, πάντα διαπιστώνουμε από τις συνομιλίες μας με τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι κακός ο συντονισμός, ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για την έκθεση δύο παρατηρήσεις τώρα, για την ε, Human Development. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι 20% της ε, βοήθειας θα πρέπει να παραμείνουν σε θέματα παιδείας και υγείας και επίσης το inclusive clause θα πρέπει να είναι, close, θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η Επιτροπή. Ο κύριος Βον Μπουργκστοφ, για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές Αξιότιμε κύριε Κατσμαρέκ, θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους σας συνεχάρισαν για το εξαιρετικό αυτό έγγραφο, όπου υπογραμμίζεται τα βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά για την μελλοντική πολιτική, που θα είναι πιο εστιασμένη στις ανάγκες των πλέον φτωχών στις χώρες εταίρους. Μιλάτε και αναφέρετε στα σημαντικά θέματα, τη σημασία της βοήθειας, τη σημασία του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο της βοήθειας αυτής και στη σημασία του να διασφαλίζεται ότι επιλύουμε με συνολικό τρόπο τις υποκείμενες αιτίες των προβλημάτων. Και ότι η προσέγγιση μας θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα που υπάρχει και που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις πτυχές που αναφέρετε εδώ πέρα και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις λύσεις και τις παρατηρήσεις σας. Στις 22 Φεβρουαρίου θα συζητηθούν τα θέματα αυτά σε επίπεδο υπουργικό και ο Επιτρόπος Πίμπαλξ ε, αντιλαμβάνεται απόλυτα τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να διορθώσω μία ημερομηνία. Είπε η Πρόεδρος ότι θα εγκρίνουμε τη νέα ανακοίνωση τον Ιούλιο. Μάλλον τον Ιούνιο θα γίνει η έγκριση αυτή. Έχουμε πραγματικά περιορισμένο χρονικό διάστημα και προσπαθούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Αν υπομονούμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο Γέννη και με την Επιτροπή σας ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κατσμάρεκ για να μας μιλήσει για ορισμένα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και ιδιαίτερα του κυρίου Μαρτίνεθ που έχει απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει η διατύπωση για την αλληλεγγύη να είναι θετική και όχι αρνητική κύριε Μαρτίνεθ. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει δηλαδή να τονίσουμε ακριβώς ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων υποστηρίζει την, πολιτική, την αναπτυξιακή πολιτική ως αναπόσπαστη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει δίκιο ο κ. Μαρτίνεθ επιμένοντας σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο και το ποσοστό χρηματοδότησης. Αυτό αυτό αναφέρεται στο έγγραφο, αλλά ίσως θα μπορούσε να γίνει πιο δυναμικά, να αναφερθεί πιο δυναμικά στο έγγραφο. Νομίζω ότι το ποσοτικό δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις αυτές και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο επιθετική πολιτική και όχι τόσο αμυντική. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε κύριε Κασμάρη και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Θα το ξανασυζητήσουμε στις 22 Μαρτίου όταν θα ακούσουμε και ορισμένους εμπειρογνώμες σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τα δάνεια. Θα αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες σε σχέση δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Μελλοντική Πολιτική στα σημεία 9 και 13. Εδώ είναι λάθος σε σχέση με το 9 και το 13. Nous avons 32 amendements. Δηλαδή δύο φορές αναφέρεται το ίδιο. Ο ίδιος τίτλος. Περνάμε στη ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλες τις κάρτες σας. Δεν τις χρειαζόμαστε, αλλά θα ήθελα να σας εκφοβήσω λιγάκι, μήπως κάποια μέρα τις χρειαστούμε. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ah λοιπόν, μελλοντική ευρωπαϊκή διεθνή πολιτική επενδύσεων, Μάσο τομέα των επενδύσεων, έκθεση Bill Newton Dunn. Έχουμε 32 τροπολογία. ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είστε έτοιμοι. Επίσης, να σηκώνετε ψηλά τα χέρια γιατί δεν είναι εύκολο. Παράγραφος 1 λοιπόν. Έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. On Allez, Ας μετρήσουμε. Εγώ νομίζω ότι κρίνεται, λέει πρόεδρος. Υπάρχει και κάποιος που αμφιβάλλει. Εγώ όχι, δεν αμφέβαλα. Αλλά ας το ελέγξουμε πάλι. Ποιοι είναι υπέρ. C'est adopté. Ah bon, il faut que je refasse. Qu'est-ce qui est contre Kata. Ah non, non, non. Donc, euh, abstention. Apochès. εγκρίνεται. Καλά το είπα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην προφορική τροπολογία. Μισό λεπτό, αλλά κάποιο επικάλυψε τον κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, το δεύτερο τμήμα τη τροπολογία αυτή ήταν σε δύο τμήματα. Ψηφίσαμε το πρώτο τμήμα, έχουμε και το δεύτερο τμήμα. Το είπατε και μόνοι σα, είναι κατά τμήματα η ψηφοφορία. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, ζητώ συγγνώμη. Τη 2 υπέρ, Κατά. Απορρίπ... Αποχές. Απορρίπτεται. Καταπίπτει η επόμενη. Λοιπόν, προφορική τροπολογία παριθμών 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, μάλλον παράγραφος 1α, τροπολογία 5, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Πάλι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται, μου λένε ότι γίνεται δεκτό, ας το εγκρίνουμε. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κύριε Γκέρνης, είχατε σηκώσει το χέρι σας ή όχι. Οκτώ ψήφοι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Είχατε δίκιο, απορρίφθηκε. Λοιπόν, τροπολογία 7 υπέρ. Οχ, πάλι ξέχασα το δεύτερο τμήμα. Συγγνώμη. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, παράγραφος 2, τροπολογία 7, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2, κατά τμήματα. Κύριε Κάτσμαρκ, είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας, κυρία Πρόεδρε, άρα καταπίπτει. Τροπολογία 8, λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Συμβιβαστική 1. Κατά τμήματα και πάλι. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δεν το ξέχασα τώρα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Καταπίπτει. Καταπίπτει. Περνάμε απευθείας στην τροπολογία 11, στην παράγραφο 4. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία θυμών 3, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, σε δύο τμήματα, όχι. Καλώς. Ξεχάστε το, καταπίπτει. Συμβιβαστική δύο κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Okay. Donc, ε, λοιπόν, εδώ έχει ζητηθεί μια προφορική τροπολογία στο δεύτερο τμήμα. και δημοσίευσε οποιοδήποτε έρμα συν και την ενδεχόμενη έλλειψη πρόοδου. Υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτή την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα με την προστίκη αυτή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά.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 Προφορική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα που πηγαίνουμε Παράγραφος 5α νέα, τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5 α ναι τροπολογια 18 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην προφορική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 όχι. Έχουν ζητήσει πράσινη χωριστή ψηφοφορία. Donc c'est un split vote, donc euh, entre... κατά τμήματα Τρία συγκεκριμένα, στην παράγραφο 6. Πρώτο τμήμα, ψήφι περ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 θα προτιμήσω να ελέγξουμε. Ποιοι είναι υπέρ πάλι παρακαλώ, σκώστε τα χέρια για την τροπολογία 26. Αλλάζετε συνέχεια γνώμη, δεν είναι εύκολο δεν έχουμε ποτέ τους ίδιους αριθμούς εδώ. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, moi 14. Ah, είστε υπέρ. Είστε υπέρ. Γιατί αν κατεβάσετε το χέρι σας. Λοιπόν, ποιοι είναι κατά παρακαλώ τώρα. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Αποχές. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 όχι. Όχι, δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 29. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο τώρα της έκθεσης. Λοιπόν, σηκώστε καλά τα χέρια. Ψήφι υπέρ παρακαλώ του συνόλου της έκθεσης, της νομοδότησης. 23, 24. 24, 24. Qu'est-ce qui est contre? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Νιούτον. Passons aux décharges. Donc, euh, Απαλλαγές. Ο κύριος Βέρμαν είναι εισηγητής. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την παράγραφο 1. Α, on block, συμφωνείτε για τις τρεις πρώτες. Ποιος είναι υπέρ των τριών πρώτων παραγράφων. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Παράγραφος 6 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά υπέρ 24. Κατά τώρα. Κατά τώρα αποχές Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Μπέρμαν. Στη συνέχεια, άλλη απαλλαγή γενικός προϋπολογισμός Μπέρμαν. Προτείνω τις δύο παραγράφους, την 1 και την 4, να τις ψηφίσουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπράβο κύριε Μπέρμαν, πολύ καλά τα καταφέρατε. Τρίτη απαλλαγή. Α, όχι, όχι. Α, του κυρίου Γκέρενς είναι αυτή η απαλλαγή. Οι ειδικέ εκθέσεις ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την απαλλαγή της Επιτροπής, παράγραφος 2, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Ξαναρχίζουμε. Υπέρ σας παρακαλώ. Να σηκώνετε καλά τα χέρια να φαίνονται, να είναι ευκρινή. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 και 9 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία, υπέρ. Κρατήστε τα χέρια ψηλά, παρακαλώ. Κύριε Μαρτίνε, τι να θεωρήσω, υπέρ ή όχι. Κατά, κατά, τώρα, κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε Γκέρενς, ε, συγχαρητήρια. Στα διάφορα υπάρχει κάτι. Προσεχή συνεδρίωση στις Βρυξέλλες, ησυχία παρακαλώ, στις 3 Μαρτίου από 9 μέχρι 12.30. Τελειώνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. coordinateurs peuvent rester. Σας παρακαλώ να παραμείνουμε συντονιστές.